Εντάξει, έχουμε την κοινή συζήτηση για τις Φιλιππίνες με τρεις ε, συστάσεις του κυρίου, ε, της εκθέσης του κυρίου Μπρόκ μάλλον, συγγνώμη. Δίνουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μπρόκ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόκειται να δώσουμε συνένεση, σύμφωνη γνώμη, για την ε, συμφωνία με τις Φιλιππίνες, που υπογράφηκε στις 12 Ιουλίου του 2012. Εάν λοιπόν το υπερψηφίσουμε αυτό, αύριο μια σειρά από κράτη-μέλη που έχουν ήδη ε, έχουν ήδη κυρώσει και έτσι μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία φέτος το πρωτόκολλο της Κροατίας μαζί με το ψήφισμα είναι ένα άλλο σκέλος αυτής της συμφωνίας νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τις δημιουργίες μας σχέσεις είναι προς το συμφέρον όλων μας και πιστεύω ότι πρέπει να εδραιωθούν αυτές οι σχέσεις ώστε να μπορέσουν και οι Φιλιππίνες να προχωρήσουν στον δρόμο της δημοκρατίας και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και με πάνω από 100 εκατομμύρια κατοίκους. Οι Φιλιππίνες είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος για μας από την Ουτεοταλική Ασία. Είναι ένας ε, ένα μέρος των πιο σημαντικών διεθνών θαλάσσιων οδών, ιδιαίτερα των προερχομένων από την Κίνα. Και άρα είναι πολύ σημαντικό να βρούμε λύσεις που θα οδηγήσουν και σε σχέση με την αντιπαράθεσή τους αυτή να, ε, που θα βοηθήσουν σε μια ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Έχουν δηλαδή εδαφικές ε, διαφορές στην νότια Κινέζικη θάλασσα η επιθετική συμπεριφορά ως προς τα εγχώρια ύδατα της Κίνας να ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα και θα ήθελα εδώ να επαναλάβω μια έκκληση εκ μέρους όλων μας για την επίλυση αυτής της εδαφικής διαφοράς με βάση το εθνές δίκαιο, με ειρηνικό τρόπο. Και πιστεύω ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας δεν θα πρέπει να πληγεί. Καλό λοιπόν τους εταίρους και τους ενθαρρύνω να προχωρήσουν προς μια ειρηνική λύση και πιο στενή συνεργασία και σε σχέση με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Οι Φιλιππίνες είναι σημαντικός ε, παράγον και για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. Ένοπλες ε, δυνάμεις στη νότια χώρα είναι σε στενή σχέση με διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες όπως η Αλ-Κάιντα και η ISIS και γι' αυτό θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Πιστεύω ότι η διαδικασία ειρηνευτική Μίντεναο, η συμφωνία του Μαρτίου του 2014 για μια ειρηνική ε, διαδικασία, για μια ειρηνευτική λύση πρέπει να συνεχιστεί και να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες που απαιτούνται ώστε εν τέλει να εγκριθεί ένα νέο κοινοβούλιο. Ο νέος πρόεδρος της 30 Ιουλίου να λαμβάνει καθήκοντα. Έχει διατυπώσει κάποιες απερίφραστες ε, και σκληρές δηλώσεις για μια σκληρή γραμμή στην πολιτική που γεννούν πολλές ανησυχίες ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περαιτέρω πορεία στην ε, χώρα αυτή αλλά ελπίζουμε ότι θα θελήσει να συνεχίσει την πολιτική ε, και την ειρηνευτική διαδικασία έχει ε, τις εμπορικές προτιμήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η χώρα νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα και για άλλα κράτη της ε, Νοτιοανατολικής Ασίας κράτη ΑΣΕΑΝ ώστε να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συμφωνίες και για τις συνθήκες εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα το περιβάλλον, τη χρηστή κυβέρνηση. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει και αναγνώριση του γεγονότος ότι είναι προϋπόθεση τέτοιου είδους νομοθεσία για την χορήγηση του καθεστώτος των ε, προτιμασιακών εμπορικών σχέσεων. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, αν προχωρήσει δηλαδή η σχετική νομοθεσία, θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε στο ορατό μέλλον να δώσει και καθεστώ ελεύθερων συναλλαγών στι Φιλιππίνε. Ευχαριστώ πολύ. Κούντερ, εκ μέρου τη Αντιπροέδρου, παρακαλώ. Ο κύριος Κούντερ, σα ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον Έλμαρ Μπροκ, πρόεδρε, για το κείμενό του και για την απόψινή εισήγηση συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε για το πόσο σημαντικό είναι να δυναμώσουμε, να στεριώσουμε καλά τις σχέσεις μας με τις Φιλιππίνες. Υποτιμούμε πολλές φορές τη σημασία της χώρας που είναι μακρινή αλλά σημαντικός εταίρος για την Ένωση. Έχουμε σημαντικές εμπορικές σχέσεις. Σημαντική χώρα γιατί έχει σημαντική γεωστατηγική σχέση την Ανατολική Ασία είναι περίπλοκη η κατάσταση στη χώρα προς τα μέσα και προς τα έξω ακριβώς όπως είπατε για την διαδικασία του Μιντανάου και θα πρέπει η ενευτική αυτή συμφωνία να αξιοποιηθεί και να ληφθούν και επιπλέον νομοθετικά μέτρα. Η σχέση μας με τη χώρα όπως γνωρίζετε βασίζεται σε ένα πλούσιο σχέσεις παρελθόν γιατί Υπάρχουν αμοιβαία συμφέροντα. Έχουμε την 25η επέτειο τη σύναψη εταιρική σχέση με τη χώρα φέτο και σε αυτά τα 25 χρόνια αναπτύσσεται η χώρα μας από πολλέ πτυχέ, ανάπτυξη, βοήθεια εμπόριο αλλά βέβαια και για την ασφάλεια συνεργαζόμαστε πολύ σημαντική η διαπροσωπική επαφή που υπάρχει είναι μια χώρα που εξάγει εργατική δύναμη. Και βέβαια όσον αφορά τα δικαιώματά τους, τους σεβόμαστε εδώ στην Ευρώπη. Πάντως αναφέρατε κύριε Μπρόκ και μια νέα συμφωνία που θα δώσει καινούργια όθηση στα πράγματα. Ελπίζουμε το πλαίσιο αυτό θα είναι σύγχρονο και ότι έτσι αυτή η σχέση θα εξελιχθεί περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες. ιδίω όσον αφορά τους πολιτικούς δεσμούς, η δήλωση της 11ης Μαρτίου για τις πρόσφατες εξελίξεις και επίσης η συνεχιζόμενη υποστήριξή μας για την ειρηνευτική διαδικασία του Μιντανάου είναι κάτι το οποίο θεωρείται θετικό από τις Φιλιππίνες. Οπότε η θετική κατάληξη θα δώσει δυνατότητες στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, ριζοσπαστικοποίηση. Έχουμε κάποιες ομάδες όπως το Αμπουσαγιάβ οι οποίοι δήλωσαν ότι προσχωρούν στο Ισλαμικό κράτος. Οπότε και εμείς πρέπει να συνεργαστούμε με τη χώρα με ευφιέστερο, στενότερο τρόπο για να δούμε πώς η κυβέρνηση μπορεί αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή. Έτσι για παράδειγμα ε, όσον αφορά το ότι προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την πολιτική μας σχέση δέχτηκαν οι Φιλιππίνες να ενεργήσουν μέσω του φόρουμ του ΑΣΕΑΝ για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού. Άρα βλέπουμε ότι δεν έχουμε μόνο καταστολή, αλλά έχουμε και πρόληψη για τη ριζοψηδικοποίηση. Επίσης θα πρέπει το PCA να τεθεί σε εφαρμογή και να έχουμε και μια εμπορική συμφωνία τα αμέσω επόμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε για την εμπορική, για τη συμφωνία του ελευθέρου εμπορίου, ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συνολών και από το 2014 έχουμε τη, τη, τη ε, την ε, συνθήκη GSP Plus για τις γενικευμένες προτιμήσεις, δηλαδή το σύστημα και έτσι θα έχουμε βοήθεια όσον αφορά την ανάπτυξη και τα εργασιακά δικαιώματα. Οπότε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων Plus πρόκειται να βοηθήσει και για τις εξαγωγές της χώρας προς την Ευρώπη. Όλα αυτά σας τα παρουσιάσαμε και τον Ιανουάριο, κύριε Μπρόκ, είχατε και εσείς την έκθεση που τα είπατε. Ε, αλλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά που αναφέρεται στην απόφαση για το σίγμα γάμα πι συν ή πλάς όλα αυτά τα αναφέρετε στην έκθεσή σας γιατί αναφέρεστε στις σχετικές μεταρρυθμίσεις και σε ζητήματα όσον αφορά τις εκτελέξεις χωρίς δίκη και την ατιμορρησία. Έχουμε για το ίδιο θέμα, δηλαδή την ετοιμορρυσία, το ψήφισμά σας του 12 οι αερομεταφορές και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, σημαντικό για τη σχέση μας γιατί έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις και ελπίζουμε να υπάρξει οριζόντια συμφωνία σύντομα μεταξύ ημών και εκείνων και έχουμε βέβαια και κάποιες ε, διμερείς συμφωνίες με κάποια κράτη-μέλη. Και όλα αυτά συνάδουν με το κοινωτικό δίκαιο. Όσον αφορά τώρα την ανάπτυξη, η χώρα έχει πολλές ανισότητες, πολλά θέματα για την ανάπτυξη και όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και έχουμε το πρόγραμμα το πολιετές 14 με 20. 325 εκατομμύρια ευρώ αντιπροσωπεύει. Αυτό έχει μια μεγάλη αύξηση, σχεδόν 2,5 φορές περισσότερο από την προηγουμένη της προηγουμένης περίοδου. Άρα τώρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Φιλιππινέζικη Προεδρία του ΑΣΕΑΝ του χρόνου. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η χώρα, διότι θέλουν να στρατευτούν στο να πετύχει η συνάντηση κορυφής του ΑΣΕΑΝ. Βέβαια και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτό που είπε ο κύριος Μπροκ για τις εκλογές της 9 Μαΐου. Με πολλοί άνθρωποι κατέβηκαν να ψηφίσουν στις εκλογές και βέβαια ήταν πολύ σημαντικό και αυτό το έκανε η εκλογική επιτροπή όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ ε, η συνεργασία μάλλον με την απερχόμενη κυβέρνηση Ακουίνο και είπαμε ότι έχουμε διάφορες δηλώσεις που επικολούθησαν ε, των εκλογών και της προεκλογικής εκστρατείας και από τον νικητή αλλά και από τους άλλους. Πάντως το κράτος θέλει να επανεισάγει την θανατική ποινή. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε την ε, δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε θα συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση για τα πάντα και θα πρέπει να κρυθεί η καινούργια κυβέρνηση από το τι θα κάνει. Θα πρέπει να δούμε τις καθημερινές γραμμές της μελούσης πολιτικής και όλα αυτά θα τα δούμε και στις 15 Ιουλίου στην συνάντηση ΑΣΕΑΝ αφού το πρόεδρος αναλάβει τα καθήκοντά του. Θα έχουμε μια πλατφόρμα για θεσμικό χαρακτήρα συνεργασία με την υπογραφή της καινούργιας συμφωνίας και θα πρέπει να δούμε και, ε, τι θα γίνει και για το συμμαγεμένο προτιμήσεων και θα πώς θα προχωρήσει ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε τη συζήτηση από πλευράς των πολιτικών ομάδων. Εξ ονόματος του ΕΛΚΑ, ο κύριος Βέρνερ Λάγκεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους Προηγούμενου ομιλητέ, να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπρόκ για την εξαιρετική έκθεσή του και να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για την ανάλυση της κατάστασης. Ως πρόεδρος τη ε, αντιπροσωπείας για το ΑΣΕΑΝ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζω την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Εταιρικής σχέση και Συνεργασίας. Μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Ξέρουμε ότι στις Φιλιππίνες ε, μπορεί να άλλαξε μπορεί να γίνει αλλαγή κυβέρνηση χωρίς αιματοχυσία. Οι Φιλιππίνες έχουν υπογράψει μια σειρά δικαιωμα... Ε, συνθήκων προστασίας των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον έχουν υπογράψει μια σειρά συμφωνιών που επιτρέπει στο 65% των προϊόντων των εξαγωγών της, ε, των Φιλιππινών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην Ένωση, κάτι πετύχαμε πέρσι. Στις διαπραγματεύσεις για την η ειρήνη στο Μιντανάο. Ε, ε, εκφράσαμε την λύπη μας ότι δεν προχώρησε η υπογραφή της συμφωνίας. Ελπίζω αυτό να συμβεί με, την, με τον νέο πρόεδρο και να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της Φιλιππίνες βάσει αυτής της ε, συμφωνίας. Ευχαριστώ λοιπόν για την βοήθεια που δώσετε στο πλαίσιο αυτό για τους σοσιαλιστές. κύριος Μπετίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έγκριση τη Συμφωνία Πλαισίου Εταιρική Σχέση και Συνεργασία μεταξύ Ένωση και Φιλιππινών είναι πολύ σημαντική πράξη. Ω σκιώδη εισηγητή από του Ζελιστέ, ευχαριστώ του συναδέλφου. Ιδίω όμω ευχαριστώ τον κύριο Μπρόκ που έλαβε με μεγάλη ξυπνάδα και ισορροπία υπόψη τις τροπολογίες που προτείνουμε, επιτυχάνοντας ε, συμβιβασμούς που έτυχαν μεγάλης υποστήριξης από την Επιτροπή. Η έγκληση επιβεβαιώνει την ε, όθηση που θέλουμε να δώσουμε ως Ευρώπη στην ε, στις ελεύθερες συναλλαγές και ως ευκαιρία ανάπτυξης και της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία η συμφωνία έχει επιπλέον το ότι, σαν σημαντικό στοιχείο, το ότι αποτελεί τη βάση μιας μεγαλύτερης επέκτασης προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, που, που αναπτύσσονται πολύ περισσότερο από την Ευρώπη και έχει ε, πληθυσμούς νέους που έχουν δίψα για ζωή. Οι Φιλιππίνες είναι μια πανέμορφη χώρα με αρχαία ιστορία και παραδοσιακές σχέσεις με τη Δύση. Όπως πολλές άλλες χώρες έχει σοβαρά προβλήματα, εγκληματικότητα, διαφθορά, κατάχρηση από τις διοκτικές αρχές. πρέπει ε, να ξεχνάμε όμως ότι είναι μια μεγάλη δημοκρατία με ένα σέρμα που προασπίζεται των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προσωπικότητας. Γι' αυτό εμείς ζητάμε μια βελτίωση των δικαιωμάτων, ε, της κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλίμα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την χώρα αυτή. Τα αιτήματά μας δεν έχουν καταστρεπτικό χαρακτήρα. Ελπίζω ότι τους επόμενους μήνες η συνεργασία με τις Φιλιππίνες να προχωρήσει και στο πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο και ελπίζω ότι η νέα κυβέρνηση που εξελέγει με μεγάλη πλειοψηφία να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση. Κύριος Μπέλντερ για, ε, για το ECR. Πρόεδρε, η παράγραφος 12 του ψηφίσματος για τις ε, Φιλιππίνες εκφράζει την ανησυχία μας για τις εντάσεις που υπάρχουν στη Νότια Συνική Θάλασσα. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μα για πολλού λόγου, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, ασφάλεια της ναυσιπλοεία, κομβικό θέμα για μας. Δεύτερον, γεωπολιτική ασφάλεια. Και αυτό διακυβεύεται. Είναι σαφές ότι υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων αμφιλεγόμενων στην περιοχή της Νότιας Συνικής Θάλασσας και εμείς πρέπει να αποφύγουμε και τετελεσμένα και να υπάρξει μια διεθνής διαιτησία. Πρέπει ωστόσο, εμείς πάμε πέραν αυτών, ζητούμε να υπάρχει μια σαφής σωστή συμπεριφορά στη Νότια Συνική Θάλασσα. Δηλαδή πρέπει να επαναφέρουμε αυτό που είχαμε πει ήδη το 2002. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Άλδε, ο κύριος Κουτσούκ.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 Συνεχίστε. Όσον αφορά λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Φιλιππίνες είναι πρότυπο για την περιοχή, καθότι έχουν κυρώσει τις περισσότερες ε, συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λοιπόν ένας κατεξοχήν εταίρος μας, γι' αυτό και Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή την συμφωνία. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις Φιλιππίνες όσον αφορά την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών, τις αλλαγές του κλίματος και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Βεβαίως γνωρίζουμε τις ε, βλέψεις της Κίνας ε, για την ε, νότια Συνική θάλασσα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικρατήσει σύνεση και να προσφύγουν στο διαιτητικό δικαστήριο όσον αφορά την επίλυση των διαφορών τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2015 και πιστεύω ότι η σύναψη αυτής της συμφωνίας θα ανοίξει νέους δρόμους για τις εμπορικές συναλλαγές προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Φιλιππίνων. Για την Ενωτική Ευρωπαϊκή Ένωση ο κ. Χατζηγεωργίου. Κύριε Πρόεδρε, πάγια μας θέση είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες μπορούν να αναπτύσσουν δεσμούς εφόσον αυτό είναι προϊόν ελεύθερη βούληση των μερών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόμαστε στι Φιλιππίνε, μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα, ειδικότερα σε θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτου δικαίου και τη διαφθορά. Πολύ σοβαρέ είναι και οι εξελίξει που συμβαίνουν στη νότια Κινέζικη θάλασσα. <clears throat> Τασσόμαστε ενάντια σε μονομερεί ενέργειε που δημιουργούν εντάσει και απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα. Υποστηρίζουμε την ειρηνική επίλυση των ζητημάτων μέσα από ένα δομημένο διάλογο Στη δική μα αντίληψη, το ψήφισμα θα μπορούσε να είναι πιο ισορροπημένο, αφού αναφέρεται μόνο στην επιθετικότητα τη Κίνα και παραλείπει να αναφερθεί στις κοινέ στρατιωτικέ ασκήσει Φιλιππινών και ΗΠΑ. Τέλο, θεωρούμε προβληματική τη σύνδεση τη σημερινή συμφωνία συνεργασία με μια ενδεχόμενη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το σύνολο των χωρών τη Νοτιοανατολική Ασία πεποίθηση μα είναι ότι οι συμφωνίε ευρωπαϊκή ένωση και τρίτων κρατών θα πρέπει να έχουν στο επίκεντρό του τη βελτίωση τη θέση των πολιτών την προστασία των δικαιωμάτων του του περιβάλλοντο και την οικοδόμηση τη ειρήνη και τη σταθερότητα. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Thank you. On behalf Greens... Για τους πράσινους, ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μας στηρίζει αυτήν την συμφωνία συνεργασίας με τις Φιλιππίνες. Θεωρούμε ότι στα πλαίσια των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Φιλιππίνες θα πρέπει να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας με τη χώρα αυτή και όχι μόνο στον οικονομικό τομέα. Περιμένουμε να είναι υπεύθυνο ο, πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος των Φιλιππίνων, πιο υπεύθυνο τουλάχιστον και πιο συνετός από τις προεκλογικές του ε, δηλώσεις. Είμαστε υπέρ μιας ειρηνικής επίλυσης των εντάσεων που επικρατούν στην ε, διαφορά και σε κάθε περίπτωση θέλουμε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών. Λυπούμεθα διότι συνεχίζουν να υπάρχουν παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ε, ομάδες και οργανώσεις δεν τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζουμε ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν ε, υπογραφεί και από τις Φιλιππίνες θα τηρηθούν και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καστάλτο, μέρος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε θετικά την ιδέα να υπάρξει εταιρική συμφωνία με τις, με τις Φιλιππίνες, ακόμα και αν υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα που πρέπει να υπογραμμιστούν. Ακόμα και η χώριση του στάτου SGP Plus για τα ανθρώπινα δικαιώματα ίσως να ήταν κάπως βιαστική, λόγω όπως έχουν πει και διάφορες εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, ακόμα υπάρχουν βασανιστήρια που ασκούνται κυρίως από τις αστυνομικές αρχές, ε, τιμωρησία και απόπειρες κατά της ελευθερίας έκφρασης, ε, για να μην μιλήσουμε για τις, τους άτακτους παραστατιωτικούς, ε, τις άτακτες παραστατικές οργανώσεις. Επίσης, όσον αφορά την νότια συνική θάλασσα, υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα και λόγω της απογραφής, αν υπογραφή, η TPP. Υπάρχουν ωστόσο επίμαχα σημεία που αφορούν τις γεωπολιτικές στρατηγικές άλλων. Γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε με πραγματικά και ξεκάθαρα βήματα, όπως αυτά που υποσχέθηκε ο Πρόεδρος στην προεκλογική εκστατεία. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο. Εξ ονόματος τώρα της ομάδας ΕΝΕΦ, ο κύριος Μποργέτσιο. η κρίση μας για αυτή τη συμφωνία επηρεάζεται από τις συνέπειες που μπορεί να έχει και οι οποίες μπορεί να είναι και βλαβερές για σημαντικά κομμάτια της ευρωπαϊκής παραγωγής, κυρίως για την παραγωγή της χώρας μου της Ιταλίας. Για παράδειγμα, η συμφωνία που επιτρέπει στις Φιλιππίνες να εξάγουν χωρίς ε, φόρους το 66% το, των προϊόντων, μεταξύ των οποίων παπούτσια και άλλα, δεν ακολουθεί την ε, ε, καλή κατεύθυνση και για τις Φιλιππίνες ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, φαίνεται να θέλουν να επιτύχουν μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Όμως ούτε η σύμβαση ούτε η η συμφωνία προβλέπουν ότι σήμερα όποιος θέλει να κάνει επιχειρήσεις στις Φιλιππίνες ξεκινώντας από την Ευρώπη θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει συμφωνίες με τοπικούς ε, ε, ε, εταίρους. Και αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Ο πρόεδρος μίλησε για μεγάλα και σπουδαία σχέδια επενδυτικά, αλλά οι δικές μας μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετέχουν σε όλα αυτά. Πολύ αφιβάλλω. Ευχαριστώ κύριε Μποργέζιο. Ο κύριος Φασρίσκο Χωζέ Μίγιαν Μόνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι Φιλιππίνες είναι ένα σημαντικό μέλος της, του ΑΣΕΑΝ και μια χώρα πολύ κοντινή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κοινέ ε, ιστορικές ε, σχέσεις Πρέπει αυτή η συμφωνία να θέσει τις βάσεις για μια μεγαλύτερη διμερή συνεργασία και να τονιστεί η καταπολέμηση της στόχης, οι κλιματικές αλλαγές και η τρομοκρατία. Οι Φιλιππίνες υποφέρουν από, τον, ε, από την τρομοκρατία του Αβού Σεμφιάφ, καθώς και την, η παρουσία του ίσης είναι όλο ένα και μεγαλύτερη. Η συμφωνία πλαίσιο θα διευκολύνει τις ελεύθερες συναλλαγές ανάμεσα ε, στις ε, δύο ενότητες και με αυτό το μέσο το SPZ ε, Plus θα έχουμε καλύτερη συνεργασία. Θα πρέπει η Φιλιππίνα ωστόσο να καταπολεμήσει την παράνομη και μη δηλωμένη αλληλεία. Και τελειώνω και πάλι ε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για αυτή τη συμφωνία που διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές με αυτή τη σημαντική περιοχή του, του Ειρηνικού. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίνα Γκίλ. Καλωσορίζω την σύναψη της συμφωνίας με τις Φιλιππίνες. Είναι βάση για την ενίσχυση των σχέσεων με τη χώρα σε μια περιοχή που αποκτά γεωπολιτική σημασία. Είμαστε με, μεγάλος εταίρος της χώρας, αλλά πόσο βάρος θα έχουμε όταν το TPP τον ΙΠΑ με την περιφέρεια υλοποιηθεί, οι Φιλιππίνες το θέλουν. Αν θέλουμε να είμαστε μπροστά, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στι διαπραγματεύσει για μια συμφωνία ελεύθερου εμποδίου που θα είναι η βάση μια περιφερειακή συμφωνία με την Νοτιοανατολική Ασία. Ένα άλλο χώρο ενδιαφέρον είναι η περιοχή της Νότιας Συνικής, όπου η Κίνα ασκεί προκλήσεις σε καθημερινή βάση, απειλώντας όχι μόνο την σταθερότητα στον κόσμο αλλά και τις εμπορικές ε, οδούς που χρησιμοποιούμε. Πρέπει να βοηθήσουμε τη φίλη, να γίνουμε ε, να βοηθήσουμε την Κίνα στην ανάπτυξή της, όχι όμως αγνοώντας την, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας ανησυχεί επίσης η εκλογή του νέου Πρόεδρου. Ευχαριστώ. Ο κ. Σέινφερντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η Νοτιοανατολική Ασία, ιδίω η Νότια Συνική Θάλασσα, είναι πολύ επικίνδυνη η περιοχή. Είναι ένα hot spot στην πραγματικότητα που μπορεί να εκρηγεί οποτεδήποτε, γιατί υπάρχουν πολλές συγκρούσεις εκεί. Από την άλλη, εκεί υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό ως προς τα αρνητικά. Ε, παράλληλα στην περιοχή αναπτύσσονται και οικονομικοί τίγρεις. Είναι ζωτικό λοιπόν να έχει η Ένωση ισχυρή οικονομική και πολιτική παρουσία στην περιοχή. Οι Φιλιππίνες έχουν 100 εκατομμύρια καθολικούς πολίτες. Θέλουμε να έχουμε στενές σχέσεις και καλή επικοινωνία. Γι' αυτό καλωσορίζω την συμφωνία με τη χώρα και το γεγονός ότι θα συζητήσουμε μια συμφωνία ελεύθερου εμποδίου. Ελπίζω αυτό να γίνει γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Στρατηγικός εταίρος μας είναι οι Φιλιππίνες σε μια κρίσιμη περιοχή με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Συμφωνία συνεργασία είναι εργαλείο για να προωθήσουμε το διάλογο και να ενισχύσουμε τη συνεργασία στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και σε στρατηγικά ζητήματα. Η εταιρική σχέση και το ξεκίνημα εμπορικών διαπραγματεύσεων πρέπει να σέβεται βέβαια τις δημοκρατικές αρχές σε συμφωνία με την αρχή GSP-SYN. Αυτό θα είναι μια, φιλική, μια φυσική εξέλιξη των σχέσεων Ευρώπης-Φελπινών. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε στενές σχέσεις με όλες τις περιοχές της περιοχής. Η θετική μας θα πρέπει να έχει στόχο να δημιουργούμε έναν κοινό χώρο με κοινέ αξίες από τις οποίες θα κερδίσουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι και των δύο πλευρών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η διαδικασία eye. Πρώτος και τελευταίος, ο κ. Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η νέα εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωση Φιλιππίνων είναι σημαντική, κυρίω για τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές, οι οποίες επιχειρούν να επενδύσουν εκεί σε μια αναδυόμενη οικονομία, όπου όμως ισχύουν μισθή πείνα. Ταυτόχρονα στις Φιλιππίνες και ιδίω στα ορυχεία δεν τηρούνται βασικά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα ενώ συναντάται συχνά το φαινόμενο της παιδικής εργασίας που αφορά δύο εκατομμύρια ανηλίκους. η διαφθορά η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι ποινικέ διώξεις πολιτικών αντιπάλων είναι επίση στην ημερήσια διάταξη. οι κοινωνικές ανισότητες και οι φτώχεια στις φιλιππίνες αποτελούν λύπασμα για τους τζιχαντιστές οι οποίοι εμφανίζουν επικίνδυνη δράση. η συμφωνία εταιρικής συνεργασίας ευρωπαϊκής ένωσης φιλιππίνων όπως κάθε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με φτωχές χώρες θα πλήξει τον ευάλωτο τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη της ένωσης και θα αυξήσει την ανεργία. η ευρωπαϊκή ένωση δεν θα πρέπει στο όνομα της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών εταιριών να κλείνει τα μάτια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολύ δε περισσότερο όταν η ίδια η εταιρική σχέση δρά υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων. ευχαριστώ. την παρέμβασή και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Κέντερς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ όλους για τη σαφήνεια των παρεμβάσεών σας. Σημείωσα όλα όσα ε, προτείνετε, τις προσδοκίες σας και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την υλοποίηση αυτής της ε, συμφωνίας αλλά και όλα όσα επιθυμείτε να προσθεθούν στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των Φιλιππίνων. Βεβαίως θα συνεχίσουμε την ευάθυνση των σχέσεών μας που θα πρέπει να βασίζονται στις κοινέ μας αξίες και στα κοινά μας συμφέροντα. Μιλήσατε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το ελεύθερο εμπόριο και βεβαίως ε, την στήριξή μας στον εκδημοκρατισμό των, ε, της χώρας αυτής. Αναφερθήκατε στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά οι ανησυχίες σας δεν θα αγνοηθούν. Φυσικά και στην αξιολόγηση που κάναμε για την περίοδο από το 2014-15 και για το καθεστώς των γενικευμένων προτιμήσεων, έκθεση που υποβάλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2016 και ως προς την συμμόρφωση βάση της Σύμβασης του, των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρακολουθούμε την κατάσταση στις Φιλιππίνες και όχι μόνο παρακολουθούμε αλλά ενδυναμώνουμε και την ε, Εθνική Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν οι διεθνείς δεσμεύσεις ε, που έχουν αναλάβει οι Φιλιππίνες και βεβαίως όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις, τις εμπορικές αυτές καθεαυτές, ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2016 και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να υπογράψουμε μια πρώτη συμφωνία που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα τομέων. Ξέρετε ότι οι Φιλιππίνες ε, στην περιοχή στην οποία βρίσκονται είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος και βάσει των στοιχείων του 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στις Φιλιππίνες. Αυτό πολλές φορές το αγνοούμε στην Ευρώπη. Όλοι νομίζουμε ότι ο πρώτος εμπορικός εταίρος και επενδυτής στις Φιλιππίνες είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Όχι, είμαστε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως λοιπόν θα γίνει αξιολόγηση όσον αφορά τη βιωσιμότητα αυτών των εμπορικών σχέσεων, των οικονομικών μας σχέσεων και θα συνεχιστεί και η παρακολούθηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ε, να τα επαναλάβουμε. Βεβαίως όσον αφορά την εσωτερική και εξωτερική κατάσταση, το θέμα που αφορά την Νότια Συνική Θάλασσα, το Διαιτητικό Δικαστήριο. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι στις 11 Μαρτίου η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εμείς έχουμε περιγράψει την θέση μας για τη διατήρηση του κράτους δικαίου και για την επίλυση αυτής της διαφοράς ειρηνικά, χωρίς την χρήση βίας, και χωρίς μονομερείς επιβολές θέσεων και λύσεων. Όσον αφορά βεβαίως τα κυριαρχικά δικαιώματα, εμείς δεν έχουμε θέση και δεν παίρνουμε θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως είναι συμβαλόμενο μέρος στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης και σε κάθε περίπτωση περιμένουμε την απόφαση η οποία αναμένεται να υποβληθεί φέτος το καλοκαίρι. Τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης κατά την άποψή μας θα πρέπει να αποτελέσουν τη μοναδική λύση την μοναδική λύση που θα οδηγήσει τελικά σε επίλυση αυτής της διαφοράς. για το λαό. των ε, Φιλιππινών θεωρούμε ότι η πρόοδος αυτές τις διαπραγματεύσεις θα αποτελέσει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Εμείς στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και βεβαίως ε, οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, είναι εξαιρετικά χρονοβόρες αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα για την σταθερότητα καθώς και η υλοποίηση της Συμφωνίας ε, Οικονομικής Στήριξης της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ που ξεκίνησε ήδη από τον Αύγουστο του 2015 θα πρέπει να συνεχίσει στην υλοποίησή του. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώτη